Colleagues, can I bring the meeting to order? Λοιπόν, να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Πριν ε, ξεκινήσουμε, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ωραία. Επίσης, η έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 5ης Σεπτεμβρίου. Αντιρρήσεις. Όχι. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, καλωσορίζω μια μικρή αντιπροσωπεία της FedEx Rail, την Ευρωπαϊκή ε, Ομοσπονδία Τουριστικών και Ιστορικών Σιδηροδρόμων, εκεί στα θεωρία. Επόμενο σημείο, σημείο 3. Σχέδιο πρότασης για απόρριψη του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής ε, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 965 του 2012 για τον κανονισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις ε, πτυτικές λειτουργίες σύμφωνα με τον κανονισμό 216 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του κανονισμού. Να σας υπενθυμίσω πως αν υποστηρίζετε την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν πρέπει να ψηφίσετε ναι στην πρόταση αυτή και Εάν δεν την υποστηρίζετε, ενώ λίγης υποστηρίζετε την πρόταση της ε, Κομισιόν, ψηφίστε κατά της απόρριψης. Σαφές? Μάλιστα. Λοιπόν, να τελειώνουμε για να ανασάνουμε κιόλας. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, όχι, με συγχωρείτε. Κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο, να δούμε αν λειτουργεί. Δοκιμαστική ψηφοφορία λοιπόν. ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεν είναι κανείς πάνω από το όριο. Ωραία. Περνάμε στην κανονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κύριε σας όλοι υπέρ κατά. Υπέρ, μάλιστα. Πέρας. εγκρίνεται το αίτημα 21 εναντί 13 Να σας υπενθυμίσω αν μέσω όλης αυτής της εφορίας πως το θέμα τώρα θα πάει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είτε θα κυρωθεί είτε όχι. Απλά για να το γνωρίζετε. Δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία για το πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Να επαναλάβω, εάν, εάν η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ησυχία παρακαλώ, υποστηρίξει την θέση της Επιτροπής, τότε θα διατηρηθεί το στάτους κβό. Έτσι, για να είναι σαφές. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Περιφερειακό σήμα ποιότητας, παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης του κυρίου Ρούμπιξ. Κύριε Ρουμπίξ, αν μπορείτε να περιμένετε λίγο. Μάλιστα, έχουμε μια παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης για το περιφερειακό σήμα ποιότητας. Το λόγο έχει ο κύριος Ρούμπιξ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το περιφερειακό σήμα και η επεξεργασία του σε τοπικό επίπεδο είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η διαδικασία αυτή προωθεί την δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε δήμους ε, και περιφέρειες στον τομέα του τουρισμού. Βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών, ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό μπορούμε να δούμε τις νέες εξελίξεις και με αυτό τον ε, τρόπο βεβαίως να προωθήσουμε τις τοπικές ε, επιχειρήσεις. Και αυτό προωθεί και την ελκυστικότητα των περιφερειών ε, και συνεισφέρει στο να γίνονται πιο ενδιαφέρουσες οι περιφέρειες και βεβαίως σημασία έχει όπως είπα το σήμα αυτό της το οποίο μπορεί να συνεισφέρει στο να υπάρξουν ε, ε, δείγματα και στην πλευρά του τουρισμού και του οικοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, ποδηλατικού τουρισμού κτλ. Τέλος, θεωρώ πως ε, αυτά δεν θα πρέπει να αποτελέσουν κάτι το νέο. Υπάρχουν ήδη τέτοια ποιοτικά σήματα πρέπει να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία και να δημιουργήσουμε διακλατικά, αν θέλετε, τέτοια έργα και το σήμα αυτό της ποιότητας να αναπτυχθεί από τους ανθρώπους εκεί, επιτόπου. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μία συνεργασία για να αναπτυχθεί ο τοπικός τουρισμός να προωθήσουμε την ανταλλαγή εμπειριών και εγώ θα ήθελα να πω σε όλους τους ενδιαφερόμενους να δουν όχι μόνο τα προφοριακά μέτρα αλλά και τα μέτρα τα εκπαιδευτικά των βέλτιστων πρακτικών να υπάρξει δηλαδή αν θέλετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα και επίσης ε, για να διασφαλίσουμε την ποιότητα υπάρχουν ήδη προδιαγραφές στην Ευρώπη, π.χ. στη Γεωργία ή ονομασίες προέλευσης. Συγκεκριμένα ονόματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ιδιότητες ε, προϊόντος. Έτσι διασφαλίζεται το ότι ε, οι ιδιότητες αυτές υπάρχουν μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ε, οπότε το θέμα της, ε, τα σήματα της γεωγραφικής ε, προέλευσης δείχνουν πως πρόκειται για κάτι το ιδιαίτερο και πρέπει άρα να ανταποκρίνεται σε κάποιες προδιαγραφές. Και οι ιδιότητες αυτές βεβαίω είναι συνδεδεμένες με την κάθε περιοχή. και έτσι βεβαίως ε, διακρίνονται αυτά τα προϊόντα από άλλα προϊόντα παρόμοια αλλά όχι ίδια. Παραδοσιακά και αυτό σημαίνει πως ξέρουμε πως χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα και πως βεβαίως είναι ε, προϊόντα της παράδοσης και σχετίζονται με τις προηγούμενες γενιές. Ε, πρέπει επίσης να υπάρχουν τουλάχιστον 25 χρόνια. Αλλά Βεβαίω, εμείς από ό,τι φαίνεται στο Κοινοβούλιο θα εγκρίνουμε αυτή την πρόταση μάλλον ε, στην επόμενη θητεία. Συνεψίζοντας, θα ήθελα να πω πως ο τομέας του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της υπαίθρου. και επηρεάζει και το εισόδημα. Δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, ο τουρισμός ε, μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα από τέτοιες ε, πρωτοβουλίες, ε, μπορεί να αυξηθεί η ποιότητα, να κερδίσουν, όπως είπα, οι περιφέρειες, αυτό μπορεί να συνεισφέρει επίσης και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών, αλλά η ανάπτυξη νέων ποιοτικών ε, σημάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σημαίνει αναγκαία προσθέμενη αξία, μπορεί να οδηγήσει σε αδιαφάνεια. Αναμένω λοιπόν και την ε, συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ κύριο Σοντάντο για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου μας για την δική μας την Επιτροπή επικεντρώνει την όλη συζήτηση γύρω από τον τουρισμό. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί από μόνο του προστιθέμενη αξία σε σχέση με την αρχική πρόταση, την αρχική έκθεση. Ωστόσο θα πρέπει η γνωμοδότηση αυτή να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη συζήτηση που είχαμε εδώ στα πλαίσια της δικής μας Επιτροπής όσον αφορά το περιφερειακό σήμα ποιότητος. Θυμάστε ότι έγινε και μία δημόσια ακρόαση στην οποία είχαμε πει ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε την ποιοτική εικόνα της Ευρώπης παγκοσμίω. Δεν είμαι λοιπόν πεπισμένοι ότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο μέσω της έκθεσης αυτής και μέσω του σήματος αυτού να καταφέρουμε τελικά να πετύχουμε τον στόχο αυτό. Αν τελικά πρέπει όμως να δώσουμε ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό σήμα ποιότητος, αν πρέπει να δώσουμε ένα πιστοποιητικό τουριστικό σήμα, τότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το προϊόν αυτό τελικά θα είναι ένα προϊόν υψηλός, υψηλής ποιότητος από κάθε άποψη. Και πολύ φοβάμαι ότι η πρόταση αυτή υπολείπεται του στόχου αυτού. Πρέπει να καταβληθούν ακόμα περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ποιοτικούς τουριστικούς προορισμούς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα όχι, κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το συνάδελφό μας ε, για τη δουλειά του. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή και το νέο αυτό μέσο που προτείνεται θα βοηθήσει για την παγίωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ήπεθρο. Είναι κρίσιμη στιγμή ε, διότι ε, Έχουμε και την μεταρρύθμιση της κοινή ζωικής πολιτικής, ακούγονται διάφορα. Αυτά τα διάφορα μηνύματα ε, πιο πολύ ε, λόγω της αστάθειας ε, για την οποία γίνεται λόγος, αυτό που κάνουν να, να αποσταθεροποιούν και να ανησυχούν περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει βελτίωση, περισσότερες συνέργειες, βελτίωση της, της ποιότητας, των στοιχείων ποιότητας μεταξύ των διαφόρων κλάδων, που εμπίπτουν ε, στο πεδίο αυτό και που είναι αντικείμενο αυτού του σήματος ποιότητας. Βέβαια δεν πρέπει αυτό να οδηγήσει σε ομοιογενοποίηση, γιατί η πολυμορφία είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της υπαίθρου. Απλά οι επισκέπτες, οι τουρίστες είναι καλό να μπορούν να συγκρίνουν την ποιότητα και τις προσφορές, την προσφορά και να λαμβάνουν έτσι τις ε, αποφάσεις τους με γνώσεως. Εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών δεν θα πρέπει μόνο να δούμε τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει αυτό και στον τουρισμό αλλά και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες γιατί δεν πρέπει να χαθούν ε, οι υπηρεσίες αυτές στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το σήμα θα πρέπει να έχει και αυτή τη δυναμική. Θα ήθελα επίσης ολοκληρώνοντας να πω ότι Υπάρχει κάποιος φόβος ε, ως προς το σήμα αυτό, ότι δηλαδή ενδεχομένως θα αποδυναμώσει τις γεωγραφικές ε, ονομασίες προέλευσης. Εγώ ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να είναι ε, αβάσιμη όλη αυτή η φόβη. Πάντως έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες, γιατί έχουμε μεν το σύστημα που ισχύει μέχρι τώρα, που λειτουργεί καλά, δίνει καλά αποτελέσματα, η αναγνώριση των ευρωπαϊκών ονομασιών για τα γεωργικά προϊόντα, ένα αυτό και άλλο το νέο αυτό σύστημα Δηλαδή ένα ευρωπαϊκό σήμα, αυτό ε, είναι το ζητούμενο, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Σίγουρα αυτό ε, ο στόχο πάντω είναι ο ίδιο, δηλαδή η βελτίωση τη ανάπτυξη απασχόληση ε, στην Ήπεθρο. Thank ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εισηγητή είναι ένα θέμα δύσκολο στο Κοινοβούλιο, δύσκολο και στα κράτη-μέλη. Έχουμε κάποιες αρμοδιότητες ε, και θέλουμε να δούμε πώς θα το προωθήσουμε το θέμα. Ξέρω πως είναι πάρα πολύ επιφυλακτικά τα κράτη-μέλη γιατί λένε πως δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα και... Ε, εντάξει, σε κάποιου νομίζεις κάποιοι είναι καλύτεροι από εμά, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα περιφερειακά σήματα ποιότητας. Και κατά την άποψή μου ένα θετικό σε αυτή την πρόταση είναι πως δημιουργεί μια πλατφόρμα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών. Βλέπω κάποιες δυσκολίες σε αυτά τα οποία προτείνονται από την Κομισιόν, δηλαδή εισαγωγή ενός πιστοποιητικού ποιότητας για τον τουρισμό στην Ευρώπη. Το συζητάμε, εντάξει, έχει νόημα πράγματι να εναρμονιστεί η Ευρώπη ως ε, Ταξιδιωτικό προορισμός παγκοσμίω, αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορές. Συνολικά, ειδικά ε, η Ευρώπη στην ε, Γεωργία έχει πάρα πολύ καλέ εμπειρίε και έχει κάποιο νόημα να τις ανταλλάξουμε. Ξέρω κάποιοι που το κάνουν ήδη, π.χ. εγώ κατάγομαι από την Ήπεθρο, είμαι ε, μέλος σε μια ένωση γυναικών οι οποίες ε, συνεργάζονται πάρα πολύ ενεργά και με άλλους τοπικούς συλλόγους και με άλλα κράτη-μέλη για το τι υπάρχει ως ε, πολιτιστική παράδοση, ως τοπικά προϊόντα, την προώθησή τους κτλ. Και νομίζω πως ακριβώς αυτή η πτυχή της γνωμοδότησης είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Οπότε όπως είπα υπάρχει κάποια επιφύλαξη στα γενικά για το εάν μπορούμε να εναρμονίσουμε ε, θα είναι δύσκολο, αλλά οι ανταλλαγές είναι καλές. Και ε, βεβαίως οικοτουρισμός, ποδηλατικός τουρισμός, ε, πολιτιστική κληρονομιά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ειδικά πράγματα τα οποία υπάρχουν στην Ήπεθρο και δεν είναι τόσο γνωστά. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες ανταλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μπίσεπ από τους Πράσινους είναι εδώ. Κύριος Μένιεν. Ναι. Τώρα το, το πήρα χαμπάρι αυτό, αλλά επειδή έχω κάποια εμπειρία, νομίζω πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο. κάτι ίσω σύντομο θα μπορούσαμε να έχουμε τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια πριν γίνω βουλευτής ήμουν ε, εγώ σε ένα τοπικό συμβούλιο του Χάρτφορση, ε, μια, ένα συνεταιρισμό μεταξύ εστιατόρων και των τοπικών παραγόντων για να δημιουργήσουμε αν θέλετε ακριβώς ένα τέτοιο σήμα για την περιοχή μας, ε, για τα μικρά ξενοδοχεία που υπήρχαν, τα εστιατόρια και τα αγροκτήματα έτσι ώστε και τα εστιατόρια να σερβίρουν τοπικά προϊόντα ε, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Αλλά πέρσι βεβαίως ε, χάσαμε τη χρηματοδότηση, καταργήθηκαν αυτές οι υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης. Με αυτή την εμπειρία λοιπόν θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σούτζας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι υπέρ της ε, πρότασης ε, του σχεδίου γνωμοδότησης που μας παρουσίασε σήμερα το πρωί ο συναδελφός μας και θεωρώ ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να προχωρούμε όλο και περισσότερο σε έναν τουρισμό ο οποίος ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο στην παραγωγική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι τυχαίο αυτή τη στιγμή ότι υποβάλλουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης σε σχέση με ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τελικά την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων. Ο τουρισμός ως παραγωγική λοιπόν δραστηριότητα, ο τουρισμός ο οποίος να συνδέεται με τη γεωργία και η γεωργία η οποία με τη σειρά της γίνεται τουρισμός. Νομίζω ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να προωθήσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία και μπορούμε να τη βοηθήσουμε να διέλθει να βγει από την κρίση αυτή, ακριβώς αναπτύσσοντας τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες. Δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι αντικείμενο με την κατάσταση της παραγωγής, της δραστηριότητας, όπως βλέπουμε σε άλλους κλάδους. Το ζήτημα αυτό προφανώς, το κείμενο αυτό μπορεί ακόμα να βελτιωθεί. Μπορούμε να καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες θα αναφέρονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου αυτού. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το δίκτυο το οποίο θα συνδυάζει γεωργία και τουρισμό. Νομίζω ότι ε, σίγουρα κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε ακριβώς το είδος του τουρισμού που θέλουμε και εμείς στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μερένο. Η κυρία μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει οποιοδήποτε μέτρο έχει ως στόχο την αύξηση και τη βελτίωση της οικονομίας τουρισμού, της ανάπτυξης υπαίθρου. Πρέπει ωστόσο όμως να τονίσουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία εφίστανται αυτή τη στιγμή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καταρρύψουμε ή να διαλύσουμε όλους αυτούς τους τομείς οι οποίοι λειτουργούν σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θαρρύνουμε μια περιφερειακή συνεργασία, να υπάρχει μια καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να προωθήσουμε επίση την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά α μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε κάποια εφιστάμενα συστήματα συνεργασίες όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, όσον αφορά τον ίνο, και πολύ σύντομα θα έχουμε τέτοια δίκτυα πρόθεση ποιοτικών μη γεωργικών προϊόντων. Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν πολύ καλά. Το να δημιουργηθεί τώρα ένα νέο περιφερειακό σήμα ποιότητος, ένα νέο πιστοποιητικό ποιότητος μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση του καταναλωτή και μπορεί να βάλει κατά του υφιστάμενου συστήματο και μπορεί να αποδυναμώσει οποιαδήποτε προσπάθεια έχει καταβληθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε τα ποιοτικά προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τουρίστε και οι καταναλωτέ θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτε οι, προσ... προτάσεις που γίνονται από την γνωμοδότηση αυτή, αλλά ότι να προβλέπεται ένα νέο περιφερειακό σήμα ποιότητα, όπω σα είπα, ενδεχομένω να λειτουργήσει αρνητικά σε σχέση με τα σήματα γεωργική προέλευση που ήδη έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία άλλωστε προωθούν την ποιότητα και συνδέονται άμεσα με την περιφέρεια στην οποία παράγονται τα προϊόντα αυτά. Πρέπει να σα πω λοιπόν ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι θα πρέπει σαφώς να αναπτύξουμε περισσότερο τις ακροτικές ε, περιοχές, ότι πρέπει σαφώς να προωθήσουμε τον ακροτικό κλάδο, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ήδη ποιοτικά σήματα τα οποία υφίστανται και λειτουργούν καλά. Ας μην βάλουμε κατά των σημάτων αυτών και κατά φωτοπροσπαθειών μέσω της νέας αυτής πρότασης. Ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρούμπιξ, θέλετε να προσθέσετε κάτι atliek Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν. Ελπίζω να έχουμε καλές προτάσεις και καλή συνεργασία και σας ευχαριστώ όλους. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία κατάδεση των ανθρωπολογιών είναι η 8η Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 5 Νοεμβρίου. Άρα, κατά τροπολογιών μέχρι τις 8 Οκτωβρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών 5 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο διάταξη, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Η κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχαμε πάρα πολλές ε, τροπολογίες από διάφορες ομάδες ε, ΕΛΚ, ε, σοσιαλδημοκράτες, πράσινους και συντηρητικούς. Με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η θαλάσσια χωροταξία και οι θαλάσσιες ζώνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιτύχουμε αυτή την λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, τροπολογίες ε, πολύ επικοδομητικές ε, και πολλές θα τις ενσωματώσουμε, ικανοποιούν. Υπάρχουν πάρα πολλές που στόχο έχουν να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του τι είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο και του τι είναι πράγματι αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να παραμείνει. Αυτό ήταν και η δική μου η πρόθεση ότι δηλαδή είπα και εγώ ότι είναι μια συμφωνία πλαίσιο, είναι ένα πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται ένα πλαίσιο, αλλά να διατηρήσουν και μια ευελιξία. Ε, δεν νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Υπάρχουν τροπολογίες για το πώς θα συμβάσουμε την πλέον ανάπτυξη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πράγματι σωστό είναι το ότι ναι, θέμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες και από πλευράς οικονομικής αναπτύξης, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουμε ένα ευαίσθητο οικοσύστημα υγιές και για το μέλλον. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Επίσης, κάποιες τροπολογίες τόνισαν πως χρειαζόμαστε και τα τρία στοιχεία, δηλαδή την οικολογία, το κοινωνικό και, το, και την πτυχή του οικοσυστήματος και τα τρία αυτά βεβαίως παίζουν ένα ρόλο. Κανένα δεν πρέπει να είναι κυρίαρχο. Βεβαίω σημαντικές είναι οι διαφορετικές δομές στα κράτη-μέλη, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, συμφωνώ απολύτως. Στη Μεσόγειο έχουμε των ζητημάτων αρμοδιοτήτων για συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Επίσης διαπιστώνουμε πως η θαλάσσια χωροταξία είναι θαλάσσια χωροταξία και αυτό δεν σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να αποφασίζει για τη χωροταξία στην ξηρά. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Συμπληρώσεις είχαμε και στα άρθρα 5, 7 και 8. Εδώ πέρα πρόκειται για μια απαρίθμηση. Ήθελα απλά να ξεκαθαρίσω πως δεν είναι τελική αυτή η λίστα. Είναι ευέλικτη, μπορεί να επεκταθεί, να συμπληρωθούν πράγματα. Πρώτες ύλες, το είπα, τουρισμός, πολιτιστική κληρονομιά, συμπληρώνονται διάφορα πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες ε, και στο άρθρο 16 που αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις. Και βεβαίως μετά το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι πρέπει να λάβουμε υπόψη, ε, πώς θα τοποθετηθούμε απέναντι στην πρόταση της Κομισιόν. Γενικά θα έλεγα τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Ε, θα δω τις ε, συμβαστικές προτάσεις ήδη αυτή την εβδομάδα. Θα συναντηθώ με τους και Πώς, πώς λέγεται? Shadow meeting. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια γερμανικά. Ευχαριστώ λοιπόν Βέρνερ και στις εβδομάδες του Στρασβούργου θα έχουμε μια συνάντηση στην κάθε εβδομάδα Ολομέλειας. Θα δούμε εκεί πέρα συμβαστικές προτάσεις, οπότε ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή 5 Νοεμβρίου και σκοπεύω να συνεργαστούμε γρήγορα με τις άλλες ομάδες για να τελειώσουμε πριν το τέλος αυτής της θητείας. Εγώ καταβάλω κάθε προσπάθεια γιατί η πείρα μου είναι πως όταν ξεκινάει η νέα θητεία όλα αυτά καταλήγουν στο σιρτάρι. Και ελπίζω να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναμένω λοιπόν τα περαιτέρω σχόλιά σας. Ο κύριο Κούν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ναι, και κατέθεσε μια καλή έκθεση με την οποία συμφωνούμε σε ποσοστό 90% θα έλεγα. Έχουμε κάποιες αντιρρήσεις. Πρέπει να δούμε λίγο τα βασικά σημεία. Εμείς ασχολούμαστε με τις μεταφορές. Δηλαδή να δούμε τι θαλάσσιες συγκοινωνίες, λιμάνια και τουρισμό. Επίσης, οι γραμμές της ε, ναυτιλίας. Υπάρχει κάποια βάση ήδη εδώ πέρα, δεν πρέπει της ακτοπλοείας μάλλον. Ε, δεν πρέπει να τα ανατρέψουμε όλα εξ αρχής, πρέπει να υπάρξει βεβαίως ολοκληρωμένη διαχείριση ακτών. Βεβαίως ε, υπάρχει και ε, η κυριαρχία των κρατών, τα χωρικά τους ε, ύδατα, χώρες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωμένη διαχείριση ακτών πρέπει να το δουν το ζήτημα και πιστεύω συμφωνούμε πως ακριβώς αυτή η γαλάζια ανάπτυξη ε, που αφορά τις ακτές μας και τις θάλασσές μας είναι πάρα πολύ θετική ε, και σημαντικό ρόλο βεβαίως παίζουν και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, όταν έχουμε αιωλικά πάρκα στα ανοιχτά, στο πέλαγο, στη θάλασσα και βεβαίως πρέπει να συνοηθούμε σε κάποιους διάδρομους ε, ευρωπαϊκούς ε, για να υπάρξει μια προσθέμενη αξία και θεωρώ πως πρέπει να καθοριστούν επακριβώς και οι περιοχές ε, όπου μπορεί να υπάρξει εξόριξη διαφόρων ορυκτών και ορυκτών καυσίμων και σε σχέση με τις γειτονικές χώρες να υπάρξει μια συνεννόηση. Έχουμε κάποια δυσκολία εδώ πέρα σήμερα. Σήμερα η πλάκωσαν οι πιλότοι και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Ναι, ναι, ναι, έτσι, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας. Και, και στη θάλασσα. Και τι αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, με το Γαλιλαίο και τα λοιπά, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Νομίζω λοιπόν ε, κυρία Μάισνερ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για να έχουμε ένα συνολικό πακέτο θαλάσσιας χωροταξίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mr. Kuhn. Mr. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κούν, και τον Αλχαντράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τον Σπύρο Δανέλη και ο συγγητή τη ομάδα μου. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την εξαιρετική της δουλειά και την καλή συνεργασία που είχαμε. Εν γέννη, οι τροπολίες που έχουν κατατεθεί δείχνουν ότι στην Επιτροπή μας αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα αυτό μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για τη θαλάσσια χωροταξία στα κράτη-μέλη που ακόμη δεν ε, την ασκούν και όσα έχουν χωροτοξικό σχεδιασμό στη θάλασσα να το βελτιώσουν, να έχουν καλύτερο συντονισμό. Στόχο είναι να βελτιωθεί οδηγία. Πρώτον, ε, με διασύνδεσή τη με τους στόχους ε, ε, των ευρωπαϊκών οδηγιών για την θαλάσσια, τη συγγνώμη, ανάπτυξη, βελτίωση ε, της ε, νομοθεσίας για τη θάλασσα, της σύμβασης, της σχετικής και βέβαια θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά αν ε, το κείμενο θα, θα ήταν βελτιωμένο μετά από αυτή την πρόταση. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, για παράδειγμα. Πρέπει να θεσπιστούν κάποια μη περιβαλλοντικά κριτήρια. Εν συντομή αυτή είναι η θέση μας και εμείς στηρίζουμε την έκθεση και θα δούμε και τι συμβαστικές τροπολογίες θα προκύψουν. Κύριος Βαντάλλεν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Πράγματι έχουμε καταθέσει τροπολογίες, γιατί η πρόταση ως έχει αυτή τη στιγμή για μας είναι κάπως υπερβολική. Θεωρούμε πως τα κράτη-μέλη έχουν ένα ρόλο και πρέπει να συνεχίσουν να τον έχουν και προς τα εκεί πηγαίνουν και οι δικές μας ε, τροπολογίες. Θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο την ε, εισηγήτρια. Έχουμε καταθέσει ε, ε εισηγήτρια για ένα συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε καταθέσει τροπολογία για την αλλαγή της νομικής βάσης. Εμείς θέλουμε να έχουμε ως βάση το άρθρο 192 παράγραφος 2 για την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη χωροταξία. Θα ήθελα να το δει αυτό, σας παρακαλώ, η συγκήτρια. Μάλιστα. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Αν όχι, η κυρία Μοντέζη έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thanks. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και σας ευχαριστούμε και για τις ενδιαφέρουσες αυτές τροπολογίες που έχετε καταταθέσει. Πρέπει να σας πω ότι περισσότερες τροπολογίες βρίσκουν σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συνάδουν με το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαφώς πάρα πολλά ζητήματα δεν αντιβαίνουν στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επομένως τη βρίσκουν σύμφωνη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες δεν θα ήταν αποδεκτές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα βασικό ζήτημα είναι αυτό το οποίο μόλις υπόθηκε για την νομική βάση. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας για να επαναλάβω τα όσα λέγονται και στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν επηρεάζεται από την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο χορτεξικός σχεδιασμός των πόλεων. Υπάρχουν μόνο κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες είναι καθαρά διαδικαστικής φύσης όσον αφορά τον θαλά, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και όσον αφορά την διαχείριση των παρακτήων ζωνών, πάλι και εδώ πέρα προβλέπονται κάποιες ε, διαδικαστικοί, κάποιοι διαδικαστικοί κανονισμοί προκειμένου να προστατευθούν οι ε, παράκτιες ζώνες από αρνητικές επιπτώσεις. Επομένως, δεν μπορούμε να αναφερόμαστε στο άρθρο 192 ως νομική βάση. Δεν γίνεται καμία αναφορά σε χωροταξικό σχεδιασμό πόλεων ή υπαίθρου. Η νομική λοιπόν βάση πρέπει να συνδέεται με τον βασικό στόχο της πρότασης, το βασικό στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Ότι θέλουμε ουσιαστικά να εξυπηρετήσουμε τους στόχους της πολιτικής της γαλάζιας ανάπτυξης. Να πω επίσης ότι ακούστηκαν και κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην παράκτια διαχείριση, τη διαχείριση μάλλον των παρακτίων ζωνών και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως είπε και η συγγήτρια πολύ καλά στην παρέμβασή της και στην έκθεσή της, είναι θεμελιώδου σημασίας να λάβουμε υπόψη τη διασύνδεση αυτή και να υπάρχει πραγματικά μια διασύνδεση μεταξύ θάλασσας και στεριάς. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον και οι οποίες επηρεάζουν τις παράκτιες ζώνες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι στην πρόταση θα υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των παράκτων ζωνών. Μια διασύνδεση η οποία θα λαμβάνει υπόψη την διάδραση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στις δραστηριότητες της θάλασσας και τη στεριά. Μια ακόμη παρατήρηση αναφέρθηκε η γαλάζια ανάπτυξη από μια διαφορετική όμως οπτική γωνία. Εμείς θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους της γαλάζιας ανάπτυξης. Ας είμαστε όμως σαφείς. Ο βασικός μας στόχος είναι τα κράτη-μέλη να παραμείνουν αρμόδια για τις στρατηγικές, για το περιεχόμενο των προγραμμάτων που θα προτείνουν τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν τι θα εφαρμοστεί, πού, πότε και σε ποιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναφέρεται στις περιοχές προτεραιότητας που θα πρέπει να ισχύουν γιατί ε, η τελική αρμοδιότητα, η τελική ευθύνη όσον αφορά τις προτεραιότητες, τους χώρους προτεραιότητας βρίσκεται στα κράτη-μέλη, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασιστεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι στην πρόταση αυτή γίνεται σαφή αναφορά στι αρμοδιότητε των κρατών μελών, τα οποία είναι αρμόδια προφανώ και για τι προτεραιότητε που πρέπει να θέσουν. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ σύντομα ως αντίδραση. Για τον κύριο Φαντάλεν γιατί με ρώτησε συγκεκριμένα. Θα το δω. Πράγματι από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε εδώ πέρα με την Κομισιόν χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο θαλάσσιας χωροταξίας και πρέπει να, δει, να μπούμε και την ολοκληρωμένη διαχείριση ακτών. Κάποια κράτη-μέλη έχουν κάποιο σύστημα που λειτουργεί, δεν πρέπει να αλλάξει αυτό. Και πρέπει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κάτι να τους δώσουμε κάτι από ευρωπαϊκής ε, πλευράς ε, για να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ξέρω πως έχουν φόβους ε, τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα γίνει η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα ή χωροταξία, σε καμία περίπτωση. Χωροταξία, θαλάσσια και μη, παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Απλά θα δημιουργήσουμε εδώ πέρα ένα πλαίσιο, έτσι το βλέπω εγώ και το είδαμε και με τον κύριο Φλέγκενστάιν στο Αμβούργο. Έχουμε μια ευαισθησία ως... Ε, ε, έχει μια ευαισθησία ως καταγόμενος από το Αμβούργο που είναι λιμάνι και εκεί πέρα υπάρχει ήδη ένα καθεστώς ε, ολοκληρωμένης διαχείρισης και του λιμανιού και της αλλάς περιοχής κτλ. Οπότε δεν νομίζω πως έχουμε το δικαίωμα να έρθουμε σε σύγκρουση με τα κράτη-μέλη. Θα τα συμπεριλάβουμε για να έχουμε μια καλύτερη και βιώσιμη διαχείριση. Όπως σας είπα, θα τα ξαναπούμε αυτά και στη συζήτηση των ε, συμβαστικών τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας ε, θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. 5 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα. Ο κύριος Πάρκερ έχει έρθει. Προτείνω να κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 4 και 10 γιατί δεν έχει έρθει ούτε εισηγητής ούτε σκιώδης εισηγητές. έχει έρθει κάποιος σκιώδης. Philip's not here though, is Ο Φίλιπ όμως απουσιάζει. Mr. Zaribi isn't here. I think because the commission will give it... Και ο κύριος Ζαρίμπη λείπει. Τέσσερις και δέκα. Τέσσερις και δέκα τα ξαναλέμε. Μιλάει. Με μιλούν. Θα μας είναι το τηλεφώνο.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 Okay, colleagues. Συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο σήμερα της διάταξης. Λιμενικές υπηρεσίες. Πρώτη ανάγνωση για το σχετικό κανονισμό. Θα ακούσουμε τον κύριο Φλέκενστάιν, αλλά μετά τον κύριο Κοσίμερ, τον Επιτρόπο Περιφερειών, για τρία λεπτά, επειδή ξέρω ότι θα πρέπει να φύγει. Αν συμφωνείτε θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Πακέ, μετά στον κύριο Φλεκενστάιν και μετά στον κύριο Κασίν. Πριν τις 5 παρατέταρτο ελπίζω. Κύριε Κασίν, παρακαλώ κύριο Πάκε. Δέκα λεπτά λέει εδώ έτσι. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομος κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Νομίζω έχετε λάβει τις ε, διαφάνειες. Να σας πω καταρχάς ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ένα λιμενικό πακέτο παριθμών 3. Γνωρίζω ότι το πακέτο 1 και 2 για τους λιμένες άφησαν ζωντανές μνήμες σε πολλούς από τους ευρωβουλευτές. Δεν είναι όμως αυτό ένα τρίτο πακέτο. Ναι, και τα δακρυγόνα μας άφησε, κύριε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, η πρόταση της Κομισιόν νομίζω ότι είναι πιο ε, στοχευμένη. Λαμβάνουμε υπόψη μας κάποια από τα διδάγματα που αντλήσαμε με τις δύο πρώτες απόπειρες και γι' αυτό δίνουμε ένα νέο πλαίσιο για τους λιμένες που ε, έχουν να κάνουν με πολλούς ε, φορείς, άλλους αποτελεσματικούς, άλλους λιγότερο, διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, ένα πολύπλοκο πλαίσιο και ήταν δύσκολο λοιπόν ε, να εξασφαλίσουμε και τις υπηρεσίες, την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και τη διαφάνεια. Με αυτή την πρότασή μας λοιπόν προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την πολυπλοκότητα αφενός, αλλά και να προσθέσουμε ευρωπαϊκή αξία στους λιμένες και στις ε, δραστηριότητες του αφετέρου. Πολύ σύντομα, φαντάζομαι ότι βλέπετε στο χάρτη αυτό τα βασικά δίκτυα και αυτό τα λέει από μόνα του ουσιαστικά. Δηλαδή εξετάζουμε το θέμα και από το πρίσμα της πολιτικής για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Θα ψηφίσετε κι εσείς, αλλά και το Συμβούλιο ε, μείωσε τους αριθμούς των λιμένων από 1.200 σε ένα πιο συστηματικό αριθμό, γύρω στα 300 λιμάνια, των οποίων τα 100 είναι λιμάνια του βασικού δικτύου. Έχετε λοιπόν με αυτό το εγχείρημα ε, θαλάσσιους αλλά και ε, λιμένες εσωτερικούς, ε, εσωτερικής ε, πλοή, που είναι τα σημεία εισόδου στο σύστημα των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών. Εμείς θέλουμε αυτά τα σημεία εισόδου, σε αυτό το διευρωπαϊκό δίκτυο να είναι αποτελεσματικά ε, σε όλη ε, την ε, ακτογραμμή. Έχουμε και την στρατηγική για την ανάπτυξη, αλλά αυτό το, το γνωρίζετε. Υπάρχουν λοιπόν και νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα σε αυτή την πρόταση. Τα νομοθετικά θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ένα policy paper που συνοδεύει την πρόταση της Κομισιόν και στο οποίο σας, μάλλον αναφέρουμε γενικά τι σημαίνει στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των ε, εργαζομένων ε, στους λιμές, των λιμενεργατών και των άλλων φορέων. Ήταν νομίζω θετικές οι επιπτώσεις αυτών των διαβουλεύσεων. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος τελικά έχει ξεκινήσει η ΕΣΠΟ και τα συνδικάτα στις 23 Ιουνίου είχαν την πρώτη τους συνάντηση και στις 18 ε, Οκτωβρίου θα έχουν τη δεύτερη τους συνάντηση για να δούμε πώς μπορούν να βελτιωθούν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου αυτοί οι κανονισμοί και οι εργασιακέ σχέσει. Οι εργασιακέ σχέσει δεν ε, καλύπτονται από την πρόταση τη Κομισιόν, να διευκρινίσω εδώ. Έχουμε εστιάσει στην πρότασή μα σε δύο κυρίω πτυχέ. Τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα ε, των λιμενικών ε, δραστηριοτήτων. Και πανέρχομαι σε αυτό που είπα στην ε, αρχή της παρεμβασής μου, ότι δηλαδή οι βασικές αλλαγές από τις προτάσεις του 2001 και 2004, που ήταν τα δύο πακέτα, είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα, ίσως και είναι η σημαντικότερη αλλαγή, που δεν την έχουν ακόμη αντιληφθεί ενδεχομένω όλοι οι φορεί ακόμη και γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές για να τους εξηγήσουμε την πρόταση. Δεν έχουμε λοιπόν ένα νέο μοντέλο πρόσβασης στην αγορά. Δεν μιλάμε για άνοιγμα ε, ή απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών. Η πρόταση αυτή είναι αν θέλετε μια εργαλειοθήκη όπου τα κράτη-μέλη και τα λιμάνια μπορούν να επιλέγουν ώστε οι λιμενικές υπηρεσίες να οργανώνονται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο εσωτερικοί ε, χειριστές και φορείς εκμετάλλευσης, όταν δηλαδή το λιμάνι παρέχει αυτό τις υπηρεσίες ή άνοιγμα αγορών όταν έχει αποφασιστεί ε, να παρέχονται αλλιώ υπηρεσίες από τον ε, φορέα. Θα επανέλθω. Πρόσβαση στις εμπορευματικές, στην, υπηρεσίες των επιβατών και τις εμπορευματικές δεν καλύπτεται προς τις αγορές αυτές. Είχαμε καταλήξει ότι η πρόταση της Κομισιόν που θα εγκριθεί σύντομα για τις συμβάσεις παραχώρησης ουσιαστικά καλύπτει ε, τις πιο πολλές πτυχές. Γι' αυτό δεν ε, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συμπεριλάβουμε αυτό το κομμάτι των εμπορευματικών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι διαφανής η πρόσβαση και στην πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και η χρηματοοικονομική διαφάνεια είναι σημαντικό. Θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες και να εξασφαλίσουμε ότι οι ναυτικές υπηρεσίες, ε, η ε, διαχείριση των αποβλήτων και όλες οι άλλες υπηρεσίες θα παρέχονται πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη και μπορούν, όπως σας είπα, να διαλέξουν, να έχουν πολλές επιλογές οι φορείς. Αν έχουν όμω αυτή την τόσο μεγάλη διακριτική ευχαίρεια φορεί γιατί εμείς νομοθετούμε, ίσως είναι μια ερώτηση εύλογη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σε πολλέ περιπτώσεις υπάρχει, ε, είναι λίγο κλειστό αν θέλετε ε, το, ο κλάδο είναι κλειστό. Θέλουμε να ορίσουμε τις υπηρεσίες. Και υπάρχει και πρόβλημα με την τιμολόγηση. Ε, θέλουμε να έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο όπου όταν παρέχεται σε, από έναν πάροχο υπηρεσιών η υπηρεσία να υπάρχουν σαφείς αρχές, μια δέσμη σαφών αρχών και υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και άλλες αρχές για την τιμολόγηση. Και έπειτα να υπάρχει βέβαια έλεγχος από ένα ρυθμιστή μια ρυθμιστική αρχή. Η οικονομική ε, τώρα διαφάνεια, αυτονομία ουσιαστικά έχει να κάνει με την ε, διευκόλυνση των επενδύσεων στους ε, λιμένες, η αξιολόγηση των επιπτώσεων και παρά ότι υπήρξαν κάποιες δύσκολες χρονιές πρόσφατα με πάγωμα, μείωση των ροών, Θεωρούμε ότι οι μαζικές επενδύσεις ε, θα είναι κάτι απαραίτητο για τα λιμάνια, θα επανέλθει η κατάσταση, θα ανακάμψει και θέλουμε να διευκολύνουμε και τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Να έχουν δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και οι ιδιώτες επενδυτές για να κάνουν επενδύσεις ε, στα λιμάνια. Και αυτό θέλουμε να προσελκύσει και την επαρκή χρηματοδότηση ώστε να ε, βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τους ευρωπαϊκούς λιμένες. Τέλος, ε, θέλουμε να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και ρυθμισμένη πρόσβαση, αλλά και άλλες γενικές διατάξεις, ώστε να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες παιχνιδιού, ισότιμος ανταγωνισμός, ασφάλεια δικαίου, περισσότερες επενδύσεις, όλα αυτά ελπίζουμε να οδηγήσουν σε καλύτερο επιμορισμό των δημοσίων πόρων και σε εξοικονόμηση πόρων ε, σε βάθος χρόνου. Βέβαια προσπαθήσαμε να δούμε και ποιε θα είναι αυτές ε, οι εξοικονομήσεις. Μπορεί να είναι και δέκα δις μέχρι το 2030. Σημαντικές ε, εξοικονομήσεις λοιπόν σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξοικονομήσεις για καλύτερες υπηρεσίες μεταφόρων. Και με αυτό ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει όχι ότι θα υπάρχει απλά έτσι μια νομοθεσία ή για να έχουμε μια εστερική αγορά σε όλες τις πτυχές πολιτικής μεταφορών. Βέβαια αυτό είναι απαραίτητο, αλλά η πρόταση αποσκοπεί στο όλα τα λιμάνια της Ευρώπης να είναι αποτελεσματικές πύλες εισόδου στο ευρωπαϊκό σύστημα και να υπάρχει πλήρης αξιοποίηση όλου του συστήματος μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικτύου ευρωπαϊκών μεταφορών. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Πού είναι ο εισηγητής μας, κύριος Φλέκενστάιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Μετά την προσπάθεια των λιμενικών πακέτων 1 και 2 έχουμε το πακετάκι, το λιμενικό πακετάκι 3. Και θεωρώ πως μπορούμε να πούμε πως εδώ για πρώτη φορά έχουμε μία πρόταση η οποία αν βελτιωθεί έχει μία πιθανότητα να εγκριθεί. Δεν θέλω να εξηγήσω γιατί είναι καλύτερη. Αυτό εν μέρη έγινε όσον αφορά εμπορματικές μεταφορές, κοινωνικό διάλογο κτλ. Να αναφέρω ένα πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρος πως πρέπει να οριστεί και να συζητηθεί και ίσως δεν μπορέσατε να το δεχτείτε, αλλά είναι αυτά σημεία τα οποία θα συζητήσουμε οπωσδήποτε. Δύο προϋποθέσεις θεωρώ είναι αναγκαίες για μια λογική κατάληξη της εργασίας μας που δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόταση αυτή πρώτον. Υποθέτω πως η οδηγία παραχώρησης δικαιωμάτων όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή θα ψηφιστεί έτσι στο Κοινοβούλιο. Δεύτερον, αναμένω ή φοβάμαι, δεν ξέρω τι πρέπει να πω, την επεξεργασία της ε, οδηγίας περί κρατικών ενισχύσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού αρχές του νέου έτους και το εάν θα επιδράσει στο θέμα που συζητάμε τώρα. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε, αλλά είμαι προσεκτικός γιατί επειδή προέρχομαι από λιμάνι, ε, έχουμε καεί από το λιμενικό πακέτο 1 και 2. Θέλω να συζητήσω κάποια πράγματα. Πρώτον, το κλασικό οδηγία ή κανονισμός. Ε, κατά την άποψή μου, ε, είναι σαφές πως ε, αν έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα ο κανονισμός είναι σαφώς καλύτερος από μια οδηγία. Γιατί το χύψη πράγμα βεβαίως δεν θα πραγματοποιηθεί όπως φανταζόμαστε σε μια οδηγία. Δεύτερον, το θέμα των λιμενικών τελών όπου πρέπει να καθορίσουμε τι είναι ε, δημόσιο και δημοσιοποιείται και ποιο είναι το κομμάτι που έχει σχέση με ανταγωνισμό και δεν ε, δημοσιεύεται άρα αυτομάτως. Το τρίτο θέμα είναι οι εποπτικές αρχές και τα συμβούλια των χρηστών. Να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα του να μαζευτούν κάπου οι χρήστες ε, και να πλένε την άποψή τους, ειδικά αν δεν έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία. Και αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Όσον αφορά τώρα τις εποπτικές αρχές, οπωσδήποτε οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραπονιούνται για ένα λιμάνι, αλλά πρέπει να δούμε πραγματικά κατά πόσο ισχύει αυτό το οποίο μας είπε η Κομισιόν δηλαδή, ότι δεν θα έχουμε ένα μέγεθος ένα σύστημα για όλους, αλλά ποιες δυνατότητες ήδη υπάρχουν από σήμερα, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν και να μην χρειαστεί να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Ή τουλάχιστον να διαγράψουμε ένα φάσμα ε, εντό του οποίου θα κινηθούν αυτές οι υποπτικές αρχές. Το τέταρτο είναι το θέμα του ποιες δραστηριότητες είναι αρμοδιότητες ε, του οργανισμού λιμένος και ποιες πρέπει να αφαιθούν στην ε, αγορά. Ε, αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα οπωσδήποτε. Δηλαδή, όπου είναι θέμα ασφάλειας. Και άρα, κατά την άποψή μου, δεν είναι θέμα πρόσβασης στην αγορά και τι είναι θέμα ανταγωνισμού και πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα. Αυτό θα το δούμε προσεκτικά και δεν θα είναι απλό. Πέμπτο και τελευταίο. Σε σχέση με το άρθρο 12 θα ήταν σωστό να μπει ένας ορισμός για το τι εννοούμε υποδομή και υπερδομή. Μπορεί αυτό να μας βοηθήσει και στη λύση άλλων προβλημάτων που θα μας αποσχολήσουν του χρόνου. Θα κάνω μια πρόταση και θα το συζητήσουμε με τους σκιώδεις ηγητές να δούμε τι άποψη έχουν. Και τέλος, σε ποιο βαθμό οι ιδιωτικοί ε, λιμένες συμπεριλαμβάνονται. Αφενός, αντιλαμβάνομαι αυτούς που μου λένε δεν μπαίνουν εκεί πέρα δημόσια λεφτά, είναι δικό μας ε, το ρίσκο, το επιχειρηματικό, τι, τι δουλειά έχετε εσείς. Αλλά εάν είναι να έχουμε ε, μονοπωλιακές καταστάσεις, είναι αδιάφορο για τον χρήστη το εάν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό το λιμάνι. Οπότε δεν είναι τόσο απλή αυτή η υπόθεση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Και κάποια άλλα σημεία τα οποία δεν χρειάζεται σήμερα να τα πω. Το χρονοδιάγραμμα που μας έδωσαν εδώ πέρα είναι πολύ φιλόδοξο. 4 Νοεμβρίου λέει θα δώσω την έκθεση για μετάφραση. 5 Νοεμβρίου έχουμε μία μήνυα ακρόαση. Ευχαριστώ το Προεδρείο για το ότι το κανόνισε γιατί πρέπει να δούμε νομίζω ακριβώς πώς ένα τέτοιο κανονισμό θα επιδράσει σε λιμάνια που έχουν τελείως διαφορετική οργάνωση. Οπότε ε, δεν ξέρω αν πρέπει να έχουμε τους πάντες, ε, δηλαδή συνδικάτα, απλοηγούς ε, και τα λοιπά. Γενικά να δούμε πώς θα επιδράσει σε διαφορετικά είδη λιμανιών. Ε, χτες συναντήθηκα με εκπροσώπους από το λιμάνι του Αμβούργου, από την Κόπαρ. Ε, πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με όλους τους ε, συμμετέχοντες. Δεν χρειάζεται πιστεύω να το εξηγήσω. 3 Δεκεμβρίου μετά έχει οριστεί η προθεσμία για τις τροπολογίες. Τον Ιανουάριο θα το συζητήσουμε. Φεβρουάριο ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών και το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Είναι κρίμα το ότι η μήνυα ακρόαση θα γίνει μετά την ε, σύνταξη της έκθεσης, αλλά μπορεί πιθανώς ο εισηγητής μετά να υποβάλει ε, τροπολογίες στη δική του την έκθεση. Τέλος, θεωρώ πως έχουμε μια ευκαιρία εδώ να συζητήσουμε αυτούς τους κανόνες για να καταλήξουμε σε κάποιες βελτιώσεις και σε ένα πιθανώς ε, θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κασίμη από την Επιτροπή Περιφερειών για τρία λεπτά γιατί πρέπει να φύγετε. Μετά θα ακούσουμε τους κοιόδης ηγητές ε, πριν ακούσουμε την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Κασίμη λοιπόν για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλέκενστάιν, με τον οποίο είχα τη δυνατότητα μάλιστα να συζητήσω τα βασικά, βασικά ζητήματα, καθώς επίσης και στην Επιτροπή των Περιφερειών στις 26 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή ΚΟΤΕΡ για την Εδαφική Συνοχή, η οποία ψήφισε μία τοποθετική θέση όσον αφορά το νομικό μέσο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή οδηγία η γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Κοτέρ θα ψηφιστεί στη συνέχεια από την Ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών και σύμφωνα με την γνωμοδότηση αυτή θεωρούμε ότι ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ακραίο δεσμευτικό μέτρο, όπως ο κανονισμός δηλαδή. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε προφανώς τον κεντρικό ρόλο που έχουν τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση που συμβάλλουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Θεωρούμε λοιπόν ότι η οδηγία θα ήταν το κατάλληλο μέσο καθότι θα λάβει υπόψη του κατά αυτόν τον τρόπο τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λιμένες. Να αναφερθώ και στο ζήτημα της ασφάλειας και καθώς επίσης ε, στις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποκλειστούν ορισμένες λιμενικές υπηρεσίες από την αγορά, από την έννοια της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών. Να φέρομαι στην ε, πλοήγηση, τη ρημούλκηση και άλλες υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι λιμενικές αυτές υπηρεσίες να εξαιρεθούν και να μπορούν ουσιαστικά να εμπίπτουν περισσότερο στην εθνική νομοθεσία που υπάρχει. Επίσης, όσον αφορά το μέσο εποπτείας, το μέσο ελέγχου, Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας, το οποίο όμως και να είναι και αυτό εθνικό. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπεται ένας άλλος οργανισμός για την εποπτεία, γιατί αυτό θα δημιουργήσει και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και στο έγγραφο της Επιτροπής Κοτέρ δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον κοινωνικό διάλογο, καθώς επίσης και στο ζήτημα της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Αναγνωρίζουμε τα σημαντικά αυτά ζητήματα, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η σωστή ισορροπία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοζίμιο. Ο κύριος Γκρός έχει το λόγο. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος ο κύριος Κουμουτσάκος είναι ακόμα στην Ελλάδα και μου ζήτησε να κάνω μια εισαγωγή για λογαριασμό του. Ε, επί της αρχής χαιρετίζουμε την πρόταση της Κομισιόν αλλά και αυτά τα οποία μας είπε ήδη ο εισηγητής. Η προσέγγιση αυτή δηλαδή να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι η συνοχή με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες της Κομισιόν και για την παραχώρηση και για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι σημαντικές για εμάς γιατί ε, εδώ πέρα βεβαίως η κατάσταση έχει αλλάξει. Η Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για τις μεταφορές έχει λόγο και για τις κρατικές ενισχύσεις. Τώρα, για το θέμα κανονισμό σε οδηγία. Πάντα εμείς είμαστε υπέρ ε, του κανονισμού, γιατί τουλάχιστον έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ε, ε, όταν κάνουμε 27 διαφορετικά καθεστώτα ένα, θα είναι τουλάχιστον ένα. Αλλά, αλλά επειδή η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα, θα πρέπει να υπάρχει μία κάποια ευελιξία, αν το επιτρέπει το κείμενο και εδώ πέρα συμφωνώ με τον εισηγητή, αν το επιτρέπει να μείνουμε σε οδηγία. Το θέμα το τι μπορεί να αφαιθεί στην αγορά και τι σχετίζεται με την ασφάλεια, αυτό νομίζω το είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Εγώ μπορώ να ελπίσω μόνο το εξής, πως η συζήτηση αυτή θα γίνει με σωστές πληροφορίες να έχουμε μια αντικειμενική συζήτηση, γιατί θεωρώ πως όλες οι ομάδες θεωρούν πως η ασφάλεια δεν μπορεί να ρυθμίζεται από την αγορά, αλλά ειδικά οι πτυχές της ασφάλειας ε, απαιτούν ειδική μεταχείριση. Η διαφάνεια είναι ένα ζήτημα που συζητιέται σε πολλά λιμάνια, γι' αυτό εμείς θεωρούμε πως υποχρέωσεις διαφάνειας ειδικά εκεί όπου υπάρχει αποκλειστικός πάροχος των υπηρεσιών πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρές και χρειάζεται εκεί πέρα μια εποπτική αρχή με ισχυρή ανεξαρτησία. Κύριε συνάδελφε, κύριε Φλέκενστάιν είστε και Γερμανός και, ο... και ένας προηγούμενος ηγητής επίσης ήταν ε, από εκεί και ελπίζω μια που υπάρχει μια ενεργοποίηση αυτού του φακέλου να μπορέσετε να το ολοκληρώσετε θετικά. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Gross. Mr. De... Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκρός. Ο κύριος Ντεπάκερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να πω στον ε, κύριο Γκρός ότι υπάρχουν και κάποια βελγικά λιμάνια Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόσωπο της Κομισιόν για την παρουσίαση και τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Εμείς ε, ε, θεωρούμε καλοδεχούμε την πρόταση της Κομισιόν για τον πολύ απλό λόγο ότι γνωρίζουμε βέβαια φυσικά και την ιστορία των δύο προηγούμενων πακέτων για τα λιμάνια εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά η ώρα που πρέπει να θεσπίσουμε κοινού κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατανοούμε ότι είναι τεράστιε οι διαφορέ μεταξύ των λιμανιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά Πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι χρειαζόταν δράση, η ήπια νομοθεσία δεν αρκούσε, η μη δεσμευτική νομοθεσία. Επομένω, η πρόταση τη Κομισιόν έρχεται σε επίκαιρο, έρχεται, είναι επίκαιρη. Αυτή η προσέγγιση κατά περίπτωση δεν ήταν αρκετά διαφανής, ε, είχε πολλά κενά και θέλουμε αυτά τα κενά να τα εξαλείψουμε. Δεν θέλουμε κάθε δύο εβδομάδες να πηγαίνουμε στο δικαστήριο για να βλέπουμε αν τα πράγματα είναι καλά ή όχι. Θέλουμε να προχωρήσει πλέον αυτή η πρόταση. Ένα από τα βασικά θέματα βέβαια θα είναι η ελευθερία των ε, υπηρεσιών για τα λιμάνια. Είναι κάτι το οποίο πλέον ε, ε, το βλέπουμε γραπτό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυξηθεί ο ανταγωνισμός και θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες, αλλά θα υπάρχει και μια καλύτερη, πιο σαφής διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, ε, όπως είναι τα ευρωπαϊκά δίκτυα και άλλες υπηρεσίες. Άρα στηρίζουμε αυτή την ιδέα. Η πρόταση της Κομισιόν ε, είναι περιοριστική από αυτήν την έννοια. Αποκλείονται, εξαιρούνται πολλά πράγματα δηλαδή. Θα ήθελα να συζητήσουμε και με τους άλλους σκιώδεις ε, αυτό με το εμπαραγματικό σκέλος, δηλαδή της διακίνησης φορτίων και των υπηρεσιών ε, επιβατών. Γιατί εξαιρούνται αυτοί οι δύο τομείς. Δεν ξέρω μήπως ε, θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση που να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχει επίσης η ανάγκη ε, να περιορίσει το αριθμό των παρόχων υπηρεσιών λόγω των περιορισμών χώρου από κάποιους οργανισμούς λιμένων. Αλλά μιλήσατε και την οδηγία για τις παραχωρήσεις εσείς και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, διατάξεις που μπορεί να βοηθήσουν για να έχουμε έναν καλό ελεγκτικό μηχανισμό. Και η οικονομική διαφάνεια να κρίσιμο θέμα κατά την άποψή μου. Η έλλειψη διαφάνειας ή το γεγονός ότι είναι ε, κάπως θολά ορισμένα πράγματα, παίζονται πράγματα πίσω από κλειστές πόρτες, ε, δεν είναι κάτι καλό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα λιμενικά τέλη, φυσικά και θα πρέπει να είναι διαφανή, δεν θα είναι, πρέπει να ε, υπάρχουν διακρίσεις, αλλά υπάρχει και εμπορική λογική που ισχύει και θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εμπορική λογική. Η αυτονομία τώρα ε, των λιμενικών αρχών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις εμπορικές τους στρατηγικές, αλλά βέβαια και πάλι να υπάρχει διαφάνεια και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι θα είναι δυνατό όμως σε αυτό το πλαίσιο. για τις ε, εργασιακές σχέσεις ε, δεν υπόθηκε τίποτα. Ε, σίγουρα σεβόμαστε τον κοινωνικό διάλογο που έχει ξεκινήσει. Είναι σημαντικό, πρέπει να είναι και ανοιχτό και θέλουμε να επιτύχουμε πρόοδο στον κοινωνικό διάλογο. Αν βλέπουμε να μην προοδεύει, τότε ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε ώστε να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τις ίδιες ευκαιρίες στην αγορά. Τώρα, ότι υπάρχουν διαφορές, πράγματι, πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτό είναι σημαντικό για τα λιμάνια, αλλά και για να ευθυγραμμιστεί ο τομέας αυτός και με άλλες στρατηγικές ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό Περιμένω λοιπόν μια ανοιχτή ευρεία συζήτηση για αυτά τα διάφορα ζητήματα που έθεσα και εγώ αλλά και οι προλέσαντες συνάδελφοί μου. Ελπίζω να επιδείξουμε όλοι ανοιχτό πνεύμα για να ε, καταλήξουμε ε, σε μια πρόταση ε, που θα αφήσει στο παρελθόν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα. Κύριε Ζαρίμπη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όταν βλέπω πόσο οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν τελικά να βρίσκονται τόσο μακριά από την πραγματικότητα. 328 τα λιμάνια τα οποία εμπίπτουν στην πρόταση κανονισμού αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορες πτυχές. Πρώτον, το μέγεθος του λιμένα και το επίπεδο δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι ως προς τις πτυχές αυτές το ένα λιμάνι μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από το άλλο. Υπάρχουν ορισμένα λιμάνια που έχουν την εβδομάδα δύο-τρία σκάφη. Για παράδειγμα, στην Φιλανδία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε από την άλλη λιμένες που έχουν 600-700 σκάφη, τα οποία διέρχονται από αυτά. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο μπορούμε να έχουμε στην Ολλανδία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε κάποιους λιμένες που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, άλλους που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, άλλους λιμένες οι οποίοι συμβάλλουν στην ε, χωροταξική διαχείριση ενός ε, συγκεκριμένου χώρου, άλλοι λιμένες οι οποίοι συμβάλλουν πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία και βλέπουμε ότι από την ε, μελέτη επιπτώσεων 70% των πολιτών που βρίσκονται στους λιμένες αυτούς είναι ικανοποιημένοι από τις αποδόσεις των εν λόγω λιμένων. Πραγματικά μέσω της πρότασης αυτής θέλουμε να βελτιώσουμε ένα σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί καλά και ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά ικανοποιούμε τους ε, χρήστε των λιμένων. Εκεί που μπορώ να συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ζήτημα της διαφάνειας. Δηλαδή, πώς ε, οργανώνουμε τα τέλη τα λιμενικά. Αλλά και πάλι α δουμε πώ πώς λειτουργούν ορισμένα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι υπάρχουν εμπορικέ γενικέ συνελεύσει, οι οποίε. Ε, ουσιαστικά ανταποκρίνονται και συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Οι λιμενικοί φορείς, οι διαχειριστές των λιμένων, οι πλειοκτήτες, οι πλοηγοί. Και ξέρετε ότι με απόλυτη διαφάνεια στις γενικές αυτές συνελεύσεις καταρτίζονται τα λιμενικά τέλη. Σαφώς θα πρέπει αυτά τα τέλη στη συνέχεια να κοινοποιούνται με ένα καλύτερο τρόπο, με ένα πιο διαφανή τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί καλά. Αλλά στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μια τάση ομοιομορφίας. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εναρμόνιση αν αυτή είναι ποιοτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέτουμε ως στόχο την απόλυτη ομοιομορφία. Για παράδειγμα, όταν αφαιρόμαστε υπηρεσίες όπως η ρημούλκηση, η πλοήγηση, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι υπηρεσίε αυτές έχουν δύο βασικές προτεραιότητε. Πρώτον, η θαλάσσια ασφάλεια. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μα το επίπεδο απαιτήσεων που έχουμε πλέον σήμερα όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε ακόμα και σε τρομοκρατικέ επιθέσεις και όχι μόνο στις απλές υπηρεσίε ασφάλεια. Δεύτερον, θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε συνδικάτα πλοηγών, τα οποία πραγματικά να μπορούν να προωθούν τις επενδύσεις τις οποίες θέλουν να κάνουν στους λιμένες τους. Κατά αυτόν τον τρόπο οι λιμένες θα γίνουν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι οι λιμένες μας προφανώς δεν θα είναι ανταγωνιστικοί. Θα έχουμε ένα χαμηλό επίπεδο επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επαγγελματικών αυτών κλάδων που προφανώς θα πρέπει να διέπονται από μεγαλύτερη διαφάνεια αλλά σε καμία περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσουν έρμεο μιας άκρατης, ενός άκρατου ανταγωνισμού και νομίζω ότι και η ίδια η επίπτωση, η μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι οι ίδιοι οι χρήστε είναι ικανοποιημένοι. Μιλάμε επίση στην έκθεση αυτή για 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι το κέρδος από την επανοργάνωση που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε τι ακριβώς ανταποκρίνεται το ποσό αυτό. Δεν μας δίνονται αρκετά στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ ημών και με τα κράτη-μέλη για τις πραγματικές επενδύσεις πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές. Να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε τα δίκτυα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε καλύτερα τους λιμένες μεταξύ τους αλλά και τους λιμένες με τους άλλους τρόπους μεταφοράς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις θαλάσσιες μεταφορές και θα την καταστήσουμε και πιο ελκυστικές σε σχέση με άλλες δραστηριότητες μεταφορών. Όπως και στον σιδηροδρομικό τομέα Πιστεύω ότι ε, τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Μιλάμε για άνοιγμα των αγορών χωρί να αναφερόμαστε στι απαραίτητε επενδύσει που θα πρέπει να γίνουν στι υποδομέ προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερε επενδύσει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει κάπως την πρότασή της προκειμένου πραγματικά να αυξηθεί η διαφάνεια, να ε, λειτουργούν καλύτερα οι ρυθμιστικές αρχές, χωρίς όμως να καταστρέφουμε αυτό το οποίο ήδη ισχύει σήμερα, χωρίς να παραβλέπουμε τις πολύ καλές υποδομές που υπάρχουν σε πάρα πολλούς λιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπε και ο εισηγητής, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα αντί για κανονισμό να έχουμε οδηγία καλύτερα να πετύχουμε μια κάποια ποιοτική εναρμόνιση από το να έχουμε έναν άκαμπτο καονισμό που θα πρέπει να επιβληθεί κατά αυτόν τον τρόπο σε όλους τους λιμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Φαντάλεν, επίσης, κύριοι συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω, έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Το λόγο έχετε, κύριε Φαντάλεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα θα πω όλα μαζί. Θα πω κάποια λόγια εξ ονόματος του κύριου Μπράντμπον του ε, Σκιώδους και κάποια λόγια ε, δικά μου. Ο κύριος Μπράντμπον μου έδωσε κάποιες οδηγίες και μου είπε Ναι, θεωρεί πως δεν χρειάζεται άλλο ένα πακέτο ή πακετάκι. Έχουμε γκρίνει τα δύο λιμενικά πακέτα, δεν χρειάζονται άλλες προτάσεις και το στηρίζει αυτό με κάποια επιχειρήματα. Λέει πως η Κομισιόν τώρα μας φέρνει ένα ενιαίο πακέτο με μια ενιαία προσέγγιση η οποία δεν χρειάζεται. Ε, είναι πολύ γραφειοκρατική και γι' αυτό ο σκιώδης ηγητής ε, ε, θεωρεί και πολύ περίπλοκους τους μηχανισμούς εποπτείας και καταλήγει λέγοντας πως ε, η Κομισιόν καλό είναι να το αποσύρει ε, το πακέτο αυτό όπως εξάλλου απορρίφθηκαν και τα δύο προηγούμενα. Τώρα, αυτά από πλευράς ε, κύριου Μπραντμπορν. Εγώ έχω κάπως διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την πρότασή της. Έχουμε μια καλή προσέγγιση για την βελτίωση των λιμένων. Αυτό το οποίο δεν βλέπω είναι το πακέτο για τις κρατικές ενισχύσεις. Η οικονομική διαφάνεια πρέπει πραγματικά να υπάρχει στα λιμάνια. Εγώ στην πρόταση αυτή βλέπω πως ε, δεν έγιναν οι απαραίτητες ε, διορθώσεις. Βασικό σημείο λοιπόν οικονομική διαφάνεια χρηματικές ροές. Το άρθρο 12 εδώ πέρα έχει κρίσιμη σημασία, δεν θέλω να εξασθενήσει γιατί είναι πραγματικά πολύ βασικό σημείο. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, ε, για την θέση των πλοηγών που αναφέρονται εδώ πέρα στην ε, πρόταση αυτή. Αφενός βλέπουμε πως ε, μιλάμε για τα λιμάνια μόνο που είναι στο διευρωπαϊκό δίκτυο και στα υπόλοιπα δεν ασχολούμαστε μαζί τους, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ικανοποιεί αυτό, με Και παρόλα αυτά βλέπουμε πως η προστιθέμενη αξία των πλοηγών είναι ότι ξέρουν ακριβώς το γίνεται τοπικά, έτσι γιατί ξέρετε μετατοπίζονται οι ύφαλοι όταν είναι από άμμο και όλα αυτά. Γιατί ακριβώς η δουλειά τους κατά κύριο λόγο είναι η ασφάλεια και εγώ δεν θα ήθελα ακριβώς να εξασθενήσει καθόλου αυτό. Κατόπιν τα άρθρα 13 και 14 να είχαν απασχολήσει τότε και στο πακέτο για τα πράσινα λιμάνια και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι συμπεριλαμβάνονται εδώ πέρα. Οπότε συνολικά καλή πρόταση, έχω κάποια σημεία κριτική. θα υποβάλουμε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ κύριε Βίλσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ βεβαίω από λιμάνι προέρχομαι ενδιαφέρον ε, για την πρόταση της Κομισιόν είναι πως οι 110.000 ε, λιμενεργάτες δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Μιλάμε, λέει εδώ πέρα, θα πρέπει να διαβιλαχτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώματα σε αλλαγή επιχείρησης ε, και να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματα του υφιστάμενου προσωπικού είναι τόσο μη δεσμευτικό που σε συνδυασμό με την οδηγία παραχωρήσεων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που επίσης μας απειλεί είναι ακόμη ένα πρόβλημα για τους εργαζόμενους στα λιμάνια. Επίσης η ομάδα μου ανάλογα βλέπει και το άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού για τα δικαιώματα των εργαζομένων ως τελείως ανεπαρκές. Συνολικά δεν ξέρουμε, εμείς αμφισβητούμε την αναγκαιότητα ε, της ε, πρότασης αυτής. Ε, η Κομισιόν θεωρεί πως από Αμβέρσα μέχρι Αμβούργο στον άξονα αυτών υπάρχει ανταγωνισμός και λένε πως 80% των ερωτηθέντων θεώρησαν πως είναι ικανοποιημένοι. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μας πρέπει να διαγραφεί τελείως αυτή η πρόταση και συμφωνώ με την πρόταση της ε, Γερμανικής ε, Βουλής ε, του 1912 που είπε το εξής υπενθυμίζουμε πως κάποιες υπηρεσίες των λιμένων έχουν συμπεριληφθεί εντελώς κατά παράβαση της νομοθεσίας στην οδηγία αυτή, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες πλοήγησης ε, και άλλες. Ε, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους οι υπηρεσίες αυτής θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής οδηγίας και συμφωνώ πλήρως, αλλά εμείς είμαστε και επί της αρχής κατά αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Wells. Σας ευχαριστούμε. Βλέπω εδώ πέρα μια συνήθιστη συμμαχία που διαμορφώνεται για τους πλοηγούς, αλλά καλό είναι αυτό, καλό. Ναι. Συμβαίνουν και θαύματα. Ο κύριος Σίμονς από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή ξεκινάει τη γνωμοδότησή της με το ρητό το ότι μια του κλέφτη δυο του κλέφτη και ξέρετε τώρα είμαστε στην τρίτη φορά ήδη και είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι αντιμετωπίζει η Κομισιόν αυτό το θέμα γιατί εδώ πέρα υπάρχει η δυνατότητα να μην πειραχθεί καθόλου η διοίκηση των λιμένων. Εντάξει, να γίνει αυτό, αρκεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. και αυτό ζητάει η Επιτροπή μας. Μετά, αν συνδυάσουμε το σόφλο με την νομοθεσία, θα μπορούσαμε, με την εξάμεινη νομοθεσία θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Επίσης έχουμε και κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, που σχετίζονται με τα έξι σημεία που ανέφερε ο κύριος Φλέκενστάιν. Να ξεκινήσουμε. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως πως ε, αποκλείονται τώρα οι επιβατικές ε, και εμπορευματικές υπηρεσίες από τον ε, κανονισμό και η οριστική αξιολόγηση από τα τρία χρόνια θα πάει στα έξι χρόνια αλλά θα υπάρξει μια πρώτη έκθεση στα τρία χρόνια βεβαίως αλλά μετά θα συνεχίσει να υφίσταται ο κανονισμός τώρα για τον ε, συνδυασμό που προτείνεται. Η Επιτροπή μας θεωρεί πως ακριβώς αυτές οι λιμενικές υπηρεσίες πρέπει να είναι αντικείμενο του κανονισμού, αλλά στην εφαρμογή αυτού του κανονισμού θα πρέπει ε, πρώτα απ' όλα να ληφθούν υπόψη ε, οι πλοηγοί που πρώτος τους ρόλος είναι να συμβουλεύουν τον κυβερνήτη του κάθε πλοίου. Έτσι όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Οπότε η πτυχή της ασφάλειας κατά κύριο λόγο αφορά τους ε, πλοηγούς και άρα λέμε πως πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερος υπόψη στην εφαρμογή. Και μετά έχουμε τα ρημουλκά και τις υπόλοιπες ε, λιμενικές υπηρεσίες ε, που είναι πιο εμπορικής φύσεως. Είμαστε τελείως αντίθετοι με αυτό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 17 για ένα ανεξάρτητο εποπτικό όργανο. Είναι δουλειά της Κομισιόν να ελέγχει το εάν τα κράτη-μέλη κάνουν την δουλειά τους όσον αφορά τον έλεγχο και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Σε πάρα πολλά κράτη-μέλη ήδη ε, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση με τις επιτροπές ανταγωνισμού κτλ. τα λοιπά που εξετάζουν και τις κρατικές ενισχύσεις σε άλλα κράτη-μέλη δεν συμβαίνει ή συμβαίνει σε λιγότερο βαθμό ή εξαιρούνται τα λιμάνια εν ολίγης πρέπει να ε, υπάρξουν... Ε, πρέπει να δει η Κομισιόν το θέμα αυτό λεπτόμερο. Κύριε Σίμον, ε, αν μπορείτε συντομεύετε. Ναι, τέλος, κύριε Πρόεδρε. Στο άρθρο που αφορά τα λιμενικά τέλη, η Κομισιόν στο άρθρο 14, 1, 2 και 3 αρχίζει να έχει κάποια ελευθερία εμείς έχουμε μια πάρα πολύ απλή λύση, με μια λεξούλα που υπάρχει στη, στο άρθρο 5.5 της ανακοίνωσής μας και μετά δεν χρειάζεστε καθόλου την παράγραφο που έχετε γράψει εδώ πέρα, μπορεί να αφαιρεθεί. Σας ευχαριστώ. Τρεις έχουν μείνει και βέβαια θα ακούσουμε και τους κύριους ε, Πακέ και Φλεκενστάιν. Οι τρεις ομιλητέ, παρακαλώ να μην πέρασαν τα λεπτά. Κύριος Τούσας. το σχέδιο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη δημοσιονομική διαφάνεια των λιμένων έχει άμεση σύνδεση με τις δύο προηγούμενες προτάσεις. Κάνει μια στρατηγική επιλογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά να προχωρήσει ο βασικός της στόχος που θα της λυθούν τα χέρια έτσι ώστε να προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Με την πρότασή της στοχεύει την πλήρη απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση των λιμενικών υποδομών και των λιμενικών υπηρεσιών. Δεσπόζουσα θέση, μόνο για αυτό το πλαίσιο θα αποκτήσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που κυριαρχούν στις χερσαίες αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές που το επόμενο βήμα είναι να καθορίσουν αφού μένουν σαν θέματα εκτός του πλαισίου της πρότασης της Επιτροπής, εργασιακές σχέσεις, εμπορευματικές συναλλαγές, ζητήματα που πραγματικά ξεσήκωσαν εκατομμύρια εργαζόμενους τόσο σε ό,τι αφορά τον κλάδο αλλά και γενικότερα τους κατοίκους, όλους εμείς που ζούμε στον αστικό ιστό κοντά στα λιμάνια. Αλήθεια, γιατί κανένας μας δεν παίρνει υπόψη αυτή την αιτιολογημένη γνώμη που εμπεριέχεται, επισυνάδεται με, τα, με τις γνωμοδετήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων της Σουηδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και της Ιταλίας ότι το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία που νομοθετεί σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τις λιμενικές υποδομές και τις υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου να πω το εξή, να είμαι σύντομο να κλείσω. Υπάρχει ένας πολιτικός δογματισμός και το λέω πραγματικά με αίσθηση ευθύνη αυτό. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτόν τον ελιγμό που κάνει να είναι σίγουρη ότι δεν θα αποφύγει το επόμενο χρονικό διάστημα την αντίδραση των εργαζομένων δεν υπάρχει δηλαδή κανένας να παίρνει σοβαρά στα υπόψη του ότι υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός σήμερα που έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα το λιμάνι στον Πειραιά της Κόσκο όπου κυριαρχεί αυτός ο όμιλος και οι μεσαιωνικές σχέσεις εργασίες κυριαρχούν. Αλήθεια, γιατί οι εργαζόμενοι από τη Γαλλία, την Αγγλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία να πληρώνουν μέσα από την άμεση και έμεση φορολογία δισεκατομμύρια ευρώ για να ε, ε, κατασκευάζονται λιμενικές υποδομές στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Γερμανία και να έρχεται η Κάρνιβαλ να τις παίρνει και να τις αξιοποιεί για 99 χρόνια. Γιατί να ζούμε αυτό το μύθο, το τραγικό μύθο του Σύσυφου. Είναι μοιραίο. Όχι. Τα λιμάνια είναι στρατηγικής σημασίας τομείς και κλάδι που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και την άμυνα της χώρας. Και σε αυτό Χρειάζεται ρεαλισμός να αντιμετωπιστούν. Κυρία Γιάλα Σέντερ, σύντομα σας παρακαλώ μόνο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι όντως σύντομη. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ως προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια. Αρχικά αυτό που θέλαμε να διευθετήσουμε ήταν ε, να μην έχουμε μονοπόλια στους λιμένες. Αυτός ήταν ε, ο πρωταρχικός στόχος και αν θέλετε αυτό ήταν το εφαλτήριο για την κατάρτιση της πρότασης αυτής. Θέλαμε ουσιαστικά να πετύχουμε και έναν κάποιο βαθμό εναρμόνισης όσον αφορά τις βασικές λιμενικές υπηρεσίες και κυρίως όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες των ε, λιμενεργατών και όσον αφορά επίσης την ίδια τη διαχείριση των λιμένων. Τελικά βλέπουμε ότι τα μόνα θύματα, ε, ξυλαστήρια θύματα, που μένουν ότι δεν, δεν ε, τα βάζουμε ούτε με τις κρατικές ενισχύσεις, ούτε με τα μονοπόλια και τελικά οι επαγγελματίες του κλάδου την πληρώνουν πάλι. Αυτή είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Τι να πω, εγώ δεν συμφωνώ μια από τα ίδια, θα ήθελα να σε εξηγήσει η Κομισιόν πιο ξεκάθαρα τι αλλαγές τελικά προτείνει, τι θετικές αλλαγές προτείνει, γιατί δεν βλέπω και τίποτα διαφορετικό έχοντας ακούσει την ε, παρουσίαση. Θα εφαρμόσουμε ένα κανονισμό που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ε, και τα θύματα, επαναλαμβάνω, είναι πάλι οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού κρατικές ενισχύσεις, παραχωρήσεις, ε, λέτε ότι θα λύσει ε, η σχετική νομοθεσία ό,τι έχει να κάνει με τα λιμάνια. Τότε γιατί έχουμε αυτή την πρόταση. Κύριο Ελχαντράουι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω λέγοντας πως οπωσδήποτε είμαστε σε μια πρώτη φάση της ε, συζήτησης, αναμένουμε και την ακρόαση και τις προτάσεις του εισηγητή, αλλά θα ήθελα από τώρα να πω πως, κατά την άποψή μου, είναι θετικό το ότι η Κομισιόν δίνει το βάρος στην διαφάνεια και δεν θέλει να απελευθερώσει όλες οι υπηρεσίες όπως έκανε σε προηγούμενα πακέτα. Ελπίζω λοιπόν πως ε, δεν θα έχουμε πάλι τέτοιες προτάσεις γιατί όπως είπαν και άλλοι ομιλητές είναι ένα σύμπλεγμα σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στο οποίο πραγματικά έχει θέση ο κοινωνικός διάλογος και πρέπει να το στηρίξουμε. Και θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτό. Θα ήθελα τώρα να πω για την πρόταση πως έχουμε την εντύπωση πως ε, ε, η πρόταση είναι λίγο πάρα πολύ από οικονομική μόνο σκοπιά και θέλει να επιτρέψει εθνικές αρχές και περιφερειακές αρχές να ασχοληθούν με ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα ήταν θέμα κεντρικού κρατικού ε, σχεδιασμού, δηλαδή στον καθορισμό των υπηρεσιών και των τελών των υπηρεσιών. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια πιο εμπορική στρατηγική και να υπάρξουν διαφορές. Ε, τέλος, για το θέμα κανονισμός ή οδηγία. εξαρτάται βεβαίως και από το αποτέλεσμα της ε, συζήτησης. Καλό είναι νομίζω να αφήσουμε και στα κράτη-μέλη κάποιο περιθώριο για να προσαρμόσουν τα πράγματα στη δική τους κατάσταση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Mr. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντεπάκερ μπορεί να πάρει το λόγο. Μάλλον ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πάκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μα είδα ότι υπάρχει και μία επικοδομητική δέσμευση και συμφωνία για διάφορες πτυχές της πρότασης και ιδίω για την πτυχή της διαφάνειας. Και ακριβώς αυτό ουσιαστικά ήθελα να τονίσω όσον αφορά την πρόταση αυτή και όσον αφορά την πλοήγηση. Προφανώς θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές ροές, όσον αφορά τη διαχείριση του λιμένα και όσον αφορά τις λιμενικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική ουσία της πρότασης. Δεν πρόκειται μια πρόταση που θέλει να ανοίξει την αγορά αυτή. Η κυρία Γιάλα μας είπε ποια θα είναι η επίπτωση. Μα κοιτάξτε, η επίπτωση θα είναι ότι θα υπάρχει μια αυξημένη διαφάνεια σε αυτές τις υπηρεσίες. Και Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ισχύει αυτό και για τους πλοηγούς. Αν δείτε τη μελέτη αντικτύπου θα δείτε ότι η υπηρεσία η οποία έχει πάρει την πιο αρνητική βαθμολογία από τους χρήστες είναι η πλοήγηση. Όχι για την ποιότητά της αυτή καθ' αυτή και ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Ξέρετε ότι πολλές φορές η πλοήγηση έχει πάρει και θετικούς βαθμούς για κάποιες πτυχές. Αλλά οι χρήστες επικρίνουν την ε, σειρά με την οποία δίδεται η υπηρεσία αυτή, τη σειρά με την οποία παρέχεται, καθώς επίσης και το τέλος της εν λόγω υπηρεσίας. Θεωρούν οι χρήστες ότι η υπηρεσία δεν παρέχεται με τρόπο ιδιαίτερα ικανοποιητικό και λένε ουσιαστικά ότι θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερες εταιρείες πλοήγησης τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να επιλέξουν έναν λιμένα, μάλλον συγκεκριμένα, ένας λιμένας θα μπορούσε να επιλέξει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Επίσης οι λιμένες μπορούν να επιλέξουν να υπάρχει υποχρεωτική παροχή δημόσιας υπηρεσίας όσον αφορά την πλοήγηση. Άλλοι λιμένες θα μπορούν να επιλέξουν να ανοίξουν την αγορά της πλοήγησης. Δεν καθορίζει λοιπόν η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια τελική επιλογή θα κάνουν τα κράτη-μέλη λιμένες, αλλά προσπαθεί ουσιαστικά να φυσήσει περισσότερη διαφάνεια στην όλη διαχείριση της εν λόγω λιμενικής υπηρεσίας, καθώς επίσης και στην και στα τέλη τα οποία αντιστοιχούν σε αυτή την υπηρεσία. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα έχουμε ένα toolbox, ένα, μια εργαλειοθήκη όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιβάλλουμε ένα κοινό μοντέλο για όλους. Και προφανώς θα υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να εκφράσουν άποψή τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει σε αυτή την επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. επειδή εμένα Ήδη μου άσκησαν φοβερό λόμπινγκ οι πιλότοι των εφαίρων. Δεν θέλω να γίνει το ίδιο και με τους πλοηγούς των λιμανιών. Κύριε Φλέκενστάιν, κύριε Πρόεδρε, και μένα ε, από τη Λουφτχάνσα και, και από αλλού οι πιλότοι τις τελευταίες μέρες ε, μου άσκησαν πίεση. Τώρα, ε, για το τελικό αποτέλεσμα, εντάξει, Ελπίζω να μην θέλουμε απλά μια επιτυχία με οποιοδήποτε τίμημα. Πρέπει να λάβετε υπόψη, να αναφέρομαι στην Κομισιόν, τις διαφορές των λιμανιών. Και όταν θα κάνουμε αυτή τη μήνυα ακρόαση, νομίζω να προκύψει κάτι λογικό στο τέλος. Δεύτερον, και σημαντικό για εμένα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι ε, τόσο Προφανές το ανέφερε και ο κ. Γκρό. Το θέμα των κρατικών ισχύσεων και η οδηγία περί παραχωρήσεων δικαιωμάτων πρέπει να κινηθούν παράλληλα και να προσέξουμε να μην ε, μπουν ξανά από το παράθυρο στην συζήτηση τώρα. Για πρόσβαση στην αγορά κτλ. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε το θέμα της διαφάνειας. Ε, το θέμα του ανταγωνισμού. Εντάξει, τώρα σε κάποια επαγγέλματα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ε, αδύνατο. Αλλά οπωσδήποτε θα το δούμε αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τέλος. Να αναφερθώ στον προκατοχό μου με τον οποίο θα γευματίσω και σύντομα θα προσκαλέσω έναν δικό σας συνάδελφο, τον κύριο Ζασάδα. Θα τον ξέρετε κι εσείς. Κοιτάξτε. Ε, θα μπορούσατε νομίζω κι εσείς να πάρετε κάποιες καλές ιδέες από αυτόν. Ευχαριστώ. Very, very good. Thank you, Mr. Fleckenstein. I... Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Φλέκενστάιν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ηλικιότητα και το θάρρος, το κουράγιο. Ας είστε λοιπόν προσεκτικός όταν θα πάτε στο δείπνο αυτό που είπατε. Να επαναλάβω τα όσα είπε ο κ. Φλέκενστάιν, 5 Νοεμβρίου η μήνυα ακρόαση, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις 26 Νοεμβρίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 3η Δεκεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας το Φεβρουάριο κατά πάσα πιθανότητα και θα πάμε μάλλον στην Ολομέλεια του Μαρτίου με την έκθεση αυτή. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ όλους. Περνάμε στο επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη e-call. Κύριε Ντεμπάκερ, έχετε το λόγο. Thank you well, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πρόταση. Το έχουμε συζητήσει ε, αρκετές φορές και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί. Γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να το δούμε το ζήτημα θετικά. Όσον αφορά την εθελοντική εισαγωγή του e δεν είχε νομίζω το επιθυμητό αποτέλεσμα, οπότε η Κομισιόν έρχεται με μία πρόταση να υπάρξει υποχρέωση των κατασκευαστών να εγκαθιστούν το σύστημα αυτό στα νέα αυτοκίνητα. Και το Κοινοβούλιο ήδη είχε ζητήσει το ίδιο πράγμα. Εμείς λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικές προτάσεις. Η μία αφορά την ε, εγκατάσταση του e όταν είναι να πάρει ένα αμάξι έγκριση τύπου και το άλλο βεβαίως αφορά την εγκατάστασή του η οποία θα δίνει σήμα σε ένα κεντρικό κέντρο συναγερμού. Και βεβαίως με μεγάλη ευχαρίστηση συνεργάστηκα και με την κυρία Σενάλοβα. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Βεβαίως το σύστημα αυτό δεν μπορεί να προλάβει ατυχήματα, αλλά κερδίζει χρόνο όταν θα γίνει το ατύχημα και έτσι θα μειωθούν τα θύματα. Θα ήθελα να φερθώ σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που νομίζω πως είναι σημαντικά. Πρώτον, έχουμε την συζήτηση για το πεδίο εφαρμογής. Για τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά φορτηγά δεν νομίζω να χρειάζεται να επεκταθεί σε παλαιότερα οχήματα αυτή τη στιγμή. Επίσης θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτομάτως, να υπάρχει η δυνατότητα και χειροκίνητης ε, ενεργοποίησης και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος ε, τρόπος ε, ε, να γίνει αυτό. Όσον αφορά βεβαίως ε, το σεβασμό της ιδιωτικής ε, ζωής, θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι ενυπνώσει όπως λέμε και εδώ πέρα νομίζω πως πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση του κειμένου όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων. Επίσης στηρίζει και το σύστημα 100 12 και θα πρέπει να λειτουργεί αυτό τέλεια σε όλα τα κράτη-μέλη χωρίς ε, πρόβλημα. Και τέλος η Κομισιόν έχει καταλήξει σε μια τιμή 40 ευρώ αναεγκατάσταση, όμως οι κατασκευαστές μας λένε πως το κόστος θα είναι υψηλότερο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί για τα νούμερα τα οποία λέμε. Επίση υπάρχουν κατασκευαστέ οι οποίοι έχουν τα δικά τους εμπορικά ή ιδιωτικά συστήματα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε σχέση και με το αριθμό 112 γιατί έχουν ήδη γίνει κάποιες επενδύσεις ιδιωτικέ από πλευράς των κατασκευαστών και δεν είναι, θα πρέπει βέβαια να παραμείνει κεντρικός ο ρόλος του αριθμού 112. Θεωρώ επίσης πως το 2015 είναι κάτι το εφικτό και η πιλωτική φάση νομίζω οδήγησε στο ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα για τη μετάβαση στη νέα νομοθεσία. Βεβαίω άλλα κράτη-μέλη από έχουν δουλειά μπροστά τους, αλλά νομίζω πως μπορεί να γίνει μέχρι το 2015. Θέλουμε λοιπόν να τελειώσουμε γρήγορα με αυτό το ζήτημα και προτείνουμε το εξής, να πάει η έκθεση για μετάφραση 15 Δεκάτου, τροπολογίες μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 17 Δεκεμβρίου. Αυτό προβλέπουμε. Πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Αναμένω λοιπόν τους γεωδησηγητές και την Κομισιόν και την συνεργασία που θα έχουμε και με την ΙΜΚΟ και ελπίζω να έχουμε γρήγορα και αποτελεσματικά ε, κάποια κατάληξη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκόκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Ντεμπάκερ, πάρα πολύ καλή έκθεση. Δεν χρειάζεται νομίζω να αφαιρθώ στη λειτουργία του e το συζητάμε εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια ε, υποχρεώσαμε τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι κατασκευαστές επίσης απλά χρειάζεται λοιπόν να εφαρμοστεί. Και όλοι οι οδηγοί νομίζω πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα, όχι μόνο όσοι οδηγούν πολυτελή αυτοκίνητα. Η δε ε, Κομισιόν ακολουθεί τις προτάσεις της δικές μου και της κυρίας ε, Σεναλόβα, οπότε πρέπει νομίζω να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Σημαντικό είναι πράγματι πως όλα αυτά γίνονται με βάση τα ελάχιστα δεδομένα, όπως λέγεται, προς το νούμερο 112 θα γίνεται η κλίση. Επίσης το σύστημα θα είναι ανοιχτό και έτσι και οι ιδιώτες αλλά και τρίτα μέρη έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν περισσότερα αλλά αυτό βεβαίως σημαίνει πως θα πρέπει και ο ο ε, κάτοχος του αυτοκινήτου να αποφασίσει είτε μόνο το 112 είτε το νέο σύστημα. Στην περίπτωση δεν υπάρχει το νέο σύστημα θα πρέπει να υπάρχει αυτομάτως η κλίση στο 112. Αυτό πρέπει να είναι βασικός εξοπλισμός σε κάθε καινούριο αυτοκίνητο. Νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι το 2015, τον Οκτώβριο, αν και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω πως ε, μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα τα κρατημέλη να εργάζονται από αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία... Σε πρώτα και οι μετά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Βέβαια, μιλώ σε συγκέντρια εκ μέρους της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα e-call, την έγκριση τύπου συγκεκριμένα, δεν έχω να προσθέσω και πολλά στα όσα είπανε προλαλήσαντε. Απλά να πω ότι την έκθεση ε, αυτή για την οποία συνεργαστήκαμε τον κύριο Κόχ και η οποία συγκέντρωσε τις ψήφους της πλειοψηφίας στην Ολομέλεια, με αυτή την έκθεση λοιπόν δίνουμε μια σαφή εντολή ε, στην Κομισιόν για το πώς θα, ποια μορφή θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα. Και νομίζω ότι οι προτάσεις της Κομισιόν ε, συμπίπτουν με τα αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν προσυζήτηση μείζωνα ζητήματα, ίσως κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ε, στην προθεσμία, στο χρονοδιάγραμμα, 2015 δηλαδή, να είναι προθεσμία για όλα τα είδη οχημάτων, όπως ορίζεται και στην πρόταση. Ορισμένα από τα ζητήματα έχουν ήδη αναφερθεί. Πιστεύω ότι στην ε, διάρκεια του θα προβούμε και στις σχετικές διευκρινήσεις. Ε, φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι συμφωνούν ότι με τον κ. Ντεμπάκερ θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και θα έχουμε έτσι μια δημόσια υπηρεσία, το e-call που θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών. Ελπίζω να μπορέσουμε και στην ε, παρούσα ε, κοινοβουλευτική θητεία να ολοκληρώσουμε τα σχετικά. Τώρα κύριε Αλκαντράουλη, ο πρόεδρος έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Τζίτα θα ερχόταν, νομίζω ότι πρέπει να φτάνει τώρα από το αεροδρόμιο. Ενδεχομένω να τη επιτέθηκαν κάποιοι πιλότοι, ποιος ξέρει. Πρέπει να σας πω απλώ ότι ήταν ε, μακρά η διαδικασία από το 2005 όταν ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε το σύστημα e-call και τελικά έχει γίνει τώρα δράση προτεραιότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προφανώς θα συμβάλλει στον νέο στόχο του προγράμματος δράσης οδικής ασφάλειας προκειμένου να μειωθούν οι τραυματισμοί και τα θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη προφανώς είμαστε υπέρ της πρότασης αυτής. Τώρα εξ ονόματος της Τζίτα και των, της πολιτικής ε, ομάδας, καθώς επίσης στα πλαίσια της Τραν, πρέπει να σας πω ότι η θέση μας παραμένει η ίδια ε, που είχαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ε, έκθεση πρωτοβουλίας. Θεωρούμε ότι το e-call θα πρέπει να είναι ένα δημόσιο παρεχόμενο σύστημα το οποίο να βασίζεται σε όλα, στο 112 και να παρέχεται για όλα τα οχήματα να είναι ένα σύστημα διαλειτουργικό και από την 1η Οκτωβρίου του 2015 θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλα τα οχήματα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας πούν επίσης ποια είναι τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης στην επικράτειά τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τον διαλειτουργικό χαρακτήρα του e-call, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην οδηγία για τα Εφή συστήματα μεταφορών. Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται και τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο σύστημα e-call παντού, δηλαδή η γεωγραφική κάλυψη θα πρέπει να είναι πλήρης, απόλυτη, και όλοι οι κατασκευαστές ε, οχημάτων θα πρέπει να έχουν πλέον να παράγουν οχήματα τα οποία θα μπορούν να αναγνωρίζουν το σύστημα και δεύτερον να έχουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό στο όχημα και να συμπεριλαμβάνεται και στη βασική τιμή του αυτοκινήτου, να μην θεωρείται δηλαδή οψιών. Και κατά αυτόν τον τρόπο το σύστημα e-call θα είναι ένα σύστημα απλό και προσιτό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Ονίδη, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. you, Chair. Uh, σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη της Επιτροπής σας. Κυρία Σιναλόβα, νομίζω ότι το είπε ξεκάθαρα ότι εργαζόμαστε βάσει εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ελιγμών ή απομάκρυνσης από τη βασική εντολή που μας δώσατε. Ήσασταν πάρα πολύ σαφείς ως προς τις αρχές που πρέπει να ακολουθήσουμε δημόσια υπηρεσία η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα νέα οχήματα. Καλός τεχνικός εξοπλισμός που σε καμία περίπτωση δεν θα βάλει κατά της ιδιωτικής ζωής του χρήστη. Και όντω η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατοπτρίζει όλα αυτά, όλες αυτές τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπω και σε κάθε άλλη όμω πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει περιθώριο βελτίωση επιμέρου στοιχείων. Σίγουρα θα μπορούσε να πει κανεί ότι περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν για το είδο τη πληροφορία που αυτόματα αποστέλλεται σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Επίση, περισσότερο μπορεί να συζητηθεί το, το ζήτημα τη διασύνδεση του συστήματο e-call που, όπω είπαμε, θα βρίσκεται σε κάθε νέο όχημα από τον Οκτώβριο του 2015 και του πιο πολύπλοκου συστήματος που μπορεί να υπάρχει από έναν τρίτο φορέα και θα μπορούσαν να αναπτύξουν άλλοι κατασκευαστές. Βασικά εδώ πέρα θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ανοιχτό, ευέλικτο, όχι ένα σύστημα ξεχωριστό και άκαμπτο. Και επίσης μπορούμε περισσότερο να συζητήσουμε το ζήτημα τον Κέντρο Λήψης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης και το πώς θα μπορούν τελικά τα κράτη-μέλη να έχουν τα απαραίτητα κέντρα τα οποία θα φιλτράρουν τις κλίσεις αυτές οι οποίες είτε θα αποστέλλονται αυτόματα είτε θα αποστέλλονται με το χειρονακτικό σύστημα. Θα ήθελα να σας ζητήσω επίσης να ασχοληθείτε με κάποια ζητήματα, να μην ασχοληθείτε μάλλον με κάποια ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν την πρόταση πιο πολύπλοκη, όπως το να εξοπλιστούν αναδρομικά κάποια οχήματα. Καταλαβαίνετε ότι η τιμή θα είναι εντελώς διαφορετική στην περίπτωση αυτή. Θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, αυτόν τον αναδρομικό εξοπλισμό κάποιων οχημάτων, εφόσον το μέσο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια, Ωστόσο όμως ας μείνουμε στα πλαίσια της εντολής που μας έχει, δοθεί και ας μιλάμε ξεκάθαρα για μια δημόσια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να είναι εγκαταστημένη σε κάθε νέο όχημα. Ο κύριος Πετινέλη από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας ε, είναι αρμόδιος για, το, για την πτυχή της έγκρισης τύπου. Σας ευχαριστώ πολύ. δικιά μου Γενική Διεύθυνση ασχολείται με το σημείο 8 της ημερήσιας διαταξής σας, δηλαδή πιστοποίηση τύπου όσον αφορά την εγκατάσταση του συστήματος αυτού σε οχήματα, θα είναι υποχρεωτικό, όπως πούμε, το σύστημα αυτό για όλα τα νέα οχήματα από τον Οκτώβριο 2015 και μετά. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο από τεχνικής πλευράς και θα ήταν πάρα πολύ ακριβό να εξοπλίσουμε αναδρομικά τα παλιά οχήματα. Πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε την υποχρεωτική αυτή ημερομηνία του Οκτωβρίου 2015. Πάντως, ξέρετε, το σύστημα αυτό θα είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά, επομένω ο χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί αναδρομικά να εξοπλίσει το όχημά του. Και βέβαια το σύστημα αυτό θα είναι απόλυτα συμβατό με τον αριθμό κλήση 112. Όσον αφορά τις ερωτήσεις του εισηγητή, πρέπει να σας πω ότι το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα. Ενεργοποιείται όταν ανοίγει το iBox. Και μάλιστα όταν ενεργοποιούνται οι αερόσακοι, αυτόματα ενεργοποιείται και το σύστημα αυτό και καλεί ουσιαστικά τον αριθμό 112. Επιπλέον θα είναι υποχρεωτική η δυνατότητα της χειρονακτικής ενεργοποίησης του συστήματος. Ενδεχομένως να υπάρχει στον πίνακα οργάνων του οχήματο και ένα κόκκινο κουμπί, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να ενεργοποιεί το σύστημα αυτό. Και αυτό η επιλογή τελικά θα είναι υποχρεωτική. Επιβεβαιώνω επίσης ότι, μάλλον ο κανονισμός λέει ότι το σύστημα βρίσκεται, όπως είπαμε, εν υπνώση, λειτουργεί με έναν τρόπο λανθάνων και μπορεί ουσιαστικά να χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπηρεσίες tracking. Επίσης είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατό το σύστημα αυτό με τον αριθμό κλήσης 112 και βέβαια πρέπει να συνάδει και με τυχόν νέες υπηρεσίες που θα προτείνουν νέοι τρίτη φορείς. Ο κύριος Δεμπάκερ. Ευχαριστώ. Βλέπω πως πηγαίνουμε προς μία ε, κατεύθυνση. Από ό,τι βλέπω η συζήτηση θα αφορά μόνο το σχεδιασμό του κόκκινου κομπιού για το χειροκίνητο χειρισμό. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Η μόνη μου ερώτηση προς την γραμματεία ήταν τι γίνεται αν το τρίχρονο παιδάκι σας αποφασίσει να πατήσει το κόκκινο κουμπί. Τέλος πάντων. προθεσμία. Μάλλον, η παρουσίαση του σχέδιου έκθεση 5 Νοεμβρίου, προθεσμία για τροπολογιών 13 Νοεμβρίου, 17 Δεκεμβρίου ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια μάλλον το Φεβρουάριο. Και έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή ημερήσια διάταξη. Ήταν κάπως διαφορετική η συνάντηση ή συνεδρίασή μας σήμερα σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. 14 Οκτωβρίου, Δευτέρα, 3 με 6.30 στις Βρυξέλλες στην επόμενη συνεδρίαση. Εδώ λοιπόν λύεται η συνεδρίαση, αλλά θα αρχίσει πάρα αυτά η συνεδρίαση των συντονιστών.